υπάρχει προσέγγιση και προς τις αρχές αλλά και προς την αντιπολίτευση της χώρας αυτής. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. So, Τελειώσαμε και τη συζήτηση για την Ουκρανία. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. The first item... Το πρώτο θέμα είναι η ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Μαδαγασκάρη. Ονομαστική ψηφοφορία. Ετοιμάστε τις κάρτες σας. The joint... Θα ψηφίσουμε το κοινό σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Had the time to vote. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. And Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Ψηφοφορία 6 προτάσεων ψηφίσματος για το Γουαντάναμο και την επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής. Ψηφίζουμε το ψη... την πρόταση ψηφίσματος στο μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοινό σχέδιο ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 1 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6 παραγραφος 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 στην παραγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος. Μάλλον τροπολογία 8 παραγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτη παράγραφος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Η κυρία Βερζιά ζήτησε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη, ήθελα να παρέμβω απλώς για να ζητήσω το εξής η τροπολογία 9 να μην μπει στην παράγραφο 4 αλλά στην παράγραφο 7. Έγινε κάποιο λάθος από την πλευρά μας. Η τροπολογία 9 αφορά δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ε, και με τον τρόπο αυτό θα κατέπιπτε η άλλη τροπολογία που αφορά έτσι κι αλλιώς ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Yeah. Thank you, thank you for the Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. And 12 Ψηφίζουμε την τροπολογία 12 στην παράγραφο 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 στην παράγραφο 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για την παράγραφο 7, ψηφοφορία κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ του δεύτερου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 μετά την αιτιολογική σκέψη B. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη C έχουμε την τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G. Τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη H ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την ολοκληρωτική σκέψη H έχουμε την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη K, K, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την αιτιολογική σκέψη L τροπολογία 4 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά υπέρ ξανά κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Is Τέλος ψηφοφορία. And it's been adopted. Εγκρίνεται. Και τέλος ψηφίζουμε για την Ουκρανία πέντε προτάσεις ψηφίσματος. Ξεκινάμε με το ψήφισμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρόταση ψηφίσματος της ΓΚΟΕ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοινό ψήφισμα τριών πολιτικών ομάδων. Με ονομαστική κλίση, έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέλος, έχω να κάνω κάποιες σύντομες ανακοινώσεις στα τσαχικά. Θα τα διαβάσω λοιπόν στα τσαχικά. Θα υποβάλουμε για έγκριση τα πρακτικά πριν την επόμενη σύνοδο, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα ψηφίσματα τα οποία